el señor presidente. Buenas tardes, colega. Χαίρετε αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Άρχιε τη συνεδρία έχουν διανεμηθεί τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρία, συνεδρίας. Δεν έχει κανείς κανένα σχόλιο να κάνει στα πρακτικά. Θεωρούνται εγκεκριμένα. Σύμφωνα με τη μερίσια διάταξη, ακολουθεί η δήλωση της υπάτης εκπροσώπου της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφαλείας διπροέδρου της Επιτροπής, κυρίας Άστον, με θέμα το σεισμό στην Αιτή. Θα λάβει το λόγο επίσης ο Επίτροπος Ντεχόχτ στη συνέχεια, αλλά πρώτα η κυρία Κάθριν Άστον. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να την καλωσορίσω. Μετά από τη μακρά συνεργασία που είχαμε σε άλλους τομείς και της εύχομαι κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια των καθηκόντων σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, δηλαδή, Άστον. Uh, President, thank you very much indeed for your σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα μου επιτρέψετε να σας ενημερώσω για την κατάσταση στην Αϊτή μετά από την φρικτή τραγωδία της 12ης Ιανουαρίου.